Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση τη Επιτροπή με θέμα στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης. Ε, ο εξ της Επιτροπής το λόγο έχει ο Επίτροπος κύριος Αντόρ, Λάζλο Αντόρ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, πρέπει να βρεθεί μια στιβαρή και συστημική λύση σύντομα για την κρίση. Με σοβαρή συνέπεια αυτή τη κρίση είναι η εξαιρετικά υψηλή ανεργία. Η ανεργία η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο 10,3% στα 27 κράτη-μέλη. Ένα επίπεδο το οποίο δεν έχουμε δει από τη δεκαετία του 1990. Εντό τη Ευρωζώνη η ανεργία είναι ακόμη υψηλότερη και έχει φτάσει το 11%. Για να βρεθούν πραγματικές λύσεις στην κρίση αυτή χρειαζόμαστε μια προσέγγιση ε, με επίκεντρο της δουλειάς. Το πακέτο της απασχόλησης παρουσιάσαμε τον Απρίλιο δείχνει πως ε, οι πολιτικές απασχόλησης μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και στόχουμε ε, επίσης να εξισορροπήσουμε την οικονομική πολιτική, ενισχύοντα τον συντονισμό των πολιτικών αποσχόλη. Χρειαζόμαστε τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα δύο αυτά ζητήματα. Το πακέτο τη Κομισιόν έχει στόχο να αναπροσαρμόσει την πολιτική μα σε τρει βασικού άξονε. Πρώτα απ' όλα, στηρίζουμε τα μετραγιά, να δημιουργήσουμε δουλειέ και να αυξήσουμε τη ζήτηση εργασία σε ολόκληρη την εικόνα. Θεωρούμε την πράσινη η οικονομία, τις ε, τεχνολογίες, ε, της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και τον τομέα της υγείας, ε, τους βασικούς τομείς ε, στους οποίους θα υπάρξει ε, ανάπτυξη και βεβαίως έχουμε συγκεκριμένα σχέδια δράσης. Προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις όπως παραδείγματος χάνει υψηλότερε επιδοτήσεις για νέες δουλειές, μετάβαση των φόρων από την εργασία στο περιβάλλον που θα είναι ουδέτερη δημοσιονομικά και βεβαίως ενίσχυση των νέων επιχειρήσεων και τέλος η κοινωνική οικονομία. Δεύτερον, το πακέτο σκοπεύει να κάνει την αγορά εργασίας πιο δυναμική μέσω δίκαιων μεταρρυθμίσεων, συγκεκριμένα από απομάκρυνση εμποδίων που υπάρχουν στην κινητικότητα των εργαζομένων. Πρέπει επίσης να διευκολύνουμε τις μεταβάσεις στην αγορά εργασίας και μια πιο δυναμική ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα βοηθήσει να μειωθούν οι ανισορροπίες και ελλείψεις ε, των διαφόρων δεξιοτήτων. Γι' αυτό επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε και το πώς εξελίσσονται οι δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν σκοπεύει να βελτιώσει την κινητικότητα αφαιρώντας τα εμπόδια εκείνα που αφορούν παραδείγματο χάρη την ε, φορητότητα των συντάξεων. Επίσης θα πρέπει να βρεθεί ένα ουσιαστικό μέτρο και εργαλείο απασχόλησης ε, σε όλο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επόμενο μέτρο του πακέτου είναι να ενισχύσουμε την παρακολούθηση και την επιτήρηση των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών έτσι ώστε να μην μεν πίσω οι πολιτικές αυτές σε σχέση με τις οικονομικές πτυχές. Επίσης, σκοπεύουμε να εμπλέξουμε τους, οικονομι... τους κοινωνικούς εταίρους στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, το πακέτο αυτό ορίζει μεγαλύτερη σχέση μεταξύ των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας και των επενδύσεων από τα κοινοτικά κονδύλια και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η στήριξη του Κοινοβουλίου έχει κρίσιμη σημασία και θα μας δώσει περαιτέρω πολιτική όθηση για να αποτελέσει η απασχόληση βασικό μέρος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Ανάπτυξης. Αναμένω λοιπόν την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Τώρα ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών. Το λόγο έχει ο κύριος Ξάμπα Ρή. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρόσφατα η Κομισιόν ε, δημοσίευσε μια πρόταση για την απασχόληση. Εμείς ε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα χαιρετίζουμε αυτό το νομοθετικό πακέτο και θα στηρίξουμε αυτή την ε, πρωτοβουλία όπως το κάναμε και στην Επιτροπή Απασχόλησης στην συζήτηση για τις πρώτες αντιδράσεις στην αυτή πρότασή σας οι συνάδελφοί μου θα τονίσουν διάφορα σημεία στο πλαίσιο της συζήτησης. Θέλω και εγώ όμως να πω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζω την ρεαλιστική προσέγγιση με την οποία πλησιάζεται αυτή την νομοθετική διαδικασία. Δυστυχώς συμφωνούμε με την άποψή σας για την ανησυχητική κατάσταση στον τομέα της ανεργίας των νέων και γενικά στον τομέα της ανεργίας. Και επίσης δυστυχώς πρέπει να διαπιστώσουμε πως ε, η αξιολόγηση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων των κρατών μελών διαπιστώνει πως ε, μέχρι στιγμής οι προτάσεις των κρατών μελών δεν επαρκούν για να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Οπότε είναι καλό, θετικό το ότι η Κομισιόν επεξεργάζεται κάποιες μεσοπρόθεσμες στρατηγικές και είναι θετικό το ότι έχετε προτεραιότητες στον πράσινο τομέα, την πληροφορική, την υγεία και βεβαίως ε, χαιρετίζουμε το ότι οι φόροι που επιβαρύνουν την εργασία θα μειωθούν σύμφωνα με την πρότασή σας και βεβαίως ε, και η οδηγία για την δυνατότητα μεταφοράς ε, συνταξιδοτικών δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική και βέβαια θα πρέπει να καταρριχθούν και τα εμπόδια για τους εργαζόμενους από Βουλγαρία και Ρουμανία και σημαντικό είναι ότι ξεκινήσατε μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και οπωσδήποτε θα έχουμε και περαιτέρω συνεργασία. Μιλίες, γιατί το πρόγραμμα είναι ε, πάρα πολύ αυστηρό και ήδη έχουμε υπερβεί το χρονοδιάγραμμα εργασιών του Κοινοβουλίου. Εξ ονόματι της ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Μπέρες για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Ευρωκοινοβούλιο θέλησε να διοργανώσει αυτή τη συζήτηση με βάση το ιδέσμη για την απασχόληση που θέσατε στο τραπέζι της ε, Κομισιόν και που θεωρώ ότι είναι σημαντικό σήμερα εδώ στην ε, Σύνοδο της Ολομέλειας να το ε, πω ότι σε μια στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μιλήσει για μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη δίπλα σε όλα τα άλλα σοβαρά θέματα και σε αυτή την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη η δική σας φωνή που λέει ότι αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή. Και γι' αυτό και διοργανώσαμε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Όταν ακούμε τις προσδοκίες των Ευρωπαίων, ενώ το ποσοστό ανεργίας φτάνει σε ιστορικά ε, επίπεδα, δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά αυτό που του απασχολεί είναι να βρουν δουλειά. Και σε αυτή την προσδοκία πρέπει συγκεκριμένα να απαντήσουμε ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τους νέους η καθημερινή ζωή και οι κοινωνικές συνθήκες σκληρώνουν καθημερινά. Πώς λοιπόν να μην βλέπουμε το φάσμα μιας χαμένης γενιάς όταν ξέρουμε ότι 5,6 εκατομμύρια νέοι είναι άνεργοι και ένας στους πέντε νέους ψάχνει δουλειά και ότι η κατάσταση κινδυνεύει να μην βελτιωθεί πριν από το 2016 σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει πως κάποιο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί μέχρι ότου οι προσανατολισμοί να παράγουν αυτό το αποτέλεσμα δημιουργία απασχόληση και θα πρέπει να έχουμε τις σωστές κινήσεις. Θα πρέπει να δούμε τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης που έχουν στείλει τα κράτη-μέλη στην Κομισιόν, τελικά η δέσμευσή του να παρουσιάσουν και εθνικά σχέδια για την απασχόληση δεν ε, ακολουθήθηκε από πράξεις. Πολλοί δεν σεβάστηκαν αυτή τους τη δέσμευση. Στα σχέδια για την απασχόληση που έχετε προτείνει, εγώ θεωρώ πως δύο προτάσεις βρίσκονται στην καρδιά της συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Καταρχήν το ταμπού που εσείς άρατε ε, όσον αφορά τους ελάχιστους μισθούς. Είπατε ότι η ελάχιστη μυθή είναι ένα σημαντικό στοιχείο της συζήτηση για να καταπολεμηθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, για να καταπολεμηθεί το κοινωνικό dumping και για να τεθεί το θέμα του ε, ομαδοποιημένη ζήτηση, ε, τη εσωτερική ζήτηση, που είναι σημαντικό θέμα αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα τη έλλειψη ισορροπία, τη εσωτερική έλλειψη ισορροπία. Και έπειτα μια δεύτερη πρόταση που φαίνεται να στηρίζεται και που ξέρετε πω το Κοινοβούλιο θα σα ε, υποστηρίξει είναι η ιδέα μια εγγύηση για του νέου. Δηλαδή, ένα νέο δεν θα μπορεί να βρεθεί χωρί δουλειά, χωρί μαθητεία ή μετά από τέσσερι μήνε στην αγορά εργασία. Αυτή είναι μια πρόταση πολύ σπουδαία στην οποία αν θέλουμε πέρα από τα λόγια να προχωρήσουμε και για συγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει τις επόμενες μήνες γύρω από τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές, γύρω από τα συμπεράσματα αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προχωρήσουμε και εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας για να το καταφέρετε. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την δυναμική αυτή που πρέπει να στηρίξουμε για να προχωρήσουμε σε μια στρατηγική πέρα από τη λιτότητα που μας οδηγεί σε καταστροφή. Επόμενος ομιλητής εξ ομάδος της ε, Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ο, κύριος, ο συνάδελφος κύριος Φιλ Μπένιον, για δύο λεπτά. Uh, Αυτό το πακέτο για την απασχόληση κάνει πολλές καλοδεχούμενες ε, προτάσεις για τα κράτη-μέλη ε, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν την κρίση τα κράτη-μέλη ασχολείται με τομείς κλειδιά όπως η απασχόληση των νέων, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η κινητικότητα της εργατικής δύναμης. Και τονίζει και σε ποιους τομείς θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη πράσινη τεχνολογίας, για παράδειγμα. Ακρογωνιαίος όμως λήθος νομίζω αυτού που επιδιώκει να επιτύχει η Κομισιόν σε αυτήν την ανάκαμψη που θα δημιουργήσει θέσει εργασία είναι διαφορετικές αλλαγέ στι αγορέ εργασία. Οι αλλαγέ δεν πρέπει να γίνονται μόνο για να κάνουμε αλλαγέ. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε μελέτη επιπτώσεων. Πώ έχουν οι κανόνε τώρα για την αγορά εργασία σε κάθε κράτο μέλο και να κάνει προτάσει μεταρρύθμιση. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί φόβοι ότι αυτέ οι μεταρρυθμίσει μπορεί να βλάψουν του εργαζόμενου, να βλάψουν το κοινωνικό κράτο. Κατανοητή αυτή η φόβη, αλλά αν δεν κάνουμε τίποτα, δεν αντιμετωπίζουμε την αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων και βλέπουμε ότι πολλά κρατημέλη δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστικά. Πρέπει να είμαστε λογικοί αλλά και κοινωνικά υπεύθυνοι. Ισορροπημένες δηλαδή οι προτάσεις. Αλλά μόνο αν κάνουμε σοβαρές διορθωτικές αλλαγές τώρα μπορούμε να προωθήσουμε και να οικοδομήσουμε μια σταθερή βάση ανάπτυξης μέσω μακροπρόθεσμης βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία που να βασίζεται σε πραγματική οικονομική αποδεκτικότητα και όχι ατελείωτο το δανεισμό, θα δημιουργήσει θέσει εργασία, θα μειώσει την ανεργία. Μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία ε, μπορεί να είναι αναγκαία, δεν είναι από μόνη τη κατά ανάγκη να επαρκή. Γι' αυτό καλωσορίζω τι προτάσει που γίνονται για να αυξήσουμε την επιχειρηματικότητα, να αντιμετωπίσουμε την ενεργεια των νέων, να δώσουμε ευκαιρίε στου νέου να αναπτύξουν πολύτιμε δεξιότητε. Οι νέε επιχειρήσει είναι οι θέσει εργασία του μέλλοντο. Πρέπει να διατηρήσουμε το ρυθμό δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Πρέπει να καταργήσουμε του φραγμού για τι νέε επιχειρήσει. Η ομάδα μου των φιλελευθέρων θα συνεργαστεί μαζί σα, ε, κύριε Επίτροπε, για να προωθήσουμε αυτό το πακέτο. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο τη ομάδα των Πρασίνων τη Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, το ρόλο έχει συνάδελφο κυρία Κορνέλισεν για δύο λεπτά. Για εκατοντάδες ε, εκατομμύρια Ευρωπαίους η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η δουλειά. Οπότε θα πρέπει η πρώτη μας προτεραιότητα να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Η δήλωση αυτή είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Εμένα με ενθουσιάζει η ιδέα ενός συστήματος παρακολούθησης αγοράς εργασίας ε, για ένα σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί σε ένα εξάμεινο και βεβαίως η προσοχή που δίνεται στις πράσινες δουλειές. Εμείς το διαβάσαμε με μεγάλη ικανοποίηση. Θα μπορούσαμε να το είχαμε γράψει οι ίδιοι. 100.000 με 200.000 ε, περισσότερες θέσεις εργασίας, ε, λιγότερη χρήση καυσίμων κτλ. Αυτά νομίζω θα πρέπει να παρακινήσουν κάθε κυβέρνηση σε πράσινη πολιτική. Αλλά δεν έχω ομολόγο, μεγάλη εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή κάνει γρήγορα βήματα η Ένωσή μας προς τα εμπρός. Οικονομική, πολιτική, τραπεζική ένωση, φορολογική ένωση κτλ. Αλλά η κοινωνική πολιτική μένει πίσω. Πώς μπορούμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν βάρος και στα κοινωνικά ζητήματα. Καθώς ε, έχουν γρήγορες διαδικασίες για διάφορα ζητήματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα για να αντιμετωπιστεί η ανεργία ειδικά η ανεργία των νέων όταν χώρες ε, ακούνε να τους λένε πως ε, έχουν ε, πολύ ψηλούς μισθούς και όχι μισθούς κάτω από το όριο της φτώγειας. Αν λοιπόν να σπάνε όλα τα ταμπού, γιατί να μην σπάσουν και τα ταμπού στον κοινωνικό τομέα. Φέρτε μία οδηγία για ευρωπαϊκό ελάχιστο μισθό, φέρτε μία πρωτοβουλία για να κάνετε δεσμευτικές διάφορες ε, προτάσεις σας. Κουράγιο λοιπόν, θάρρος. Μεταρρυθμιστών, καλώ το βήμα τη συνάδελφο κυρία Μακεντάιρ για ένα λεπτό. Thank you, Mr. President. Unemployment... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανεργία είναι μεγάλη ανησυχία. Ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία. Χαιρετίζω την ανακοίνωση Τη Κομισιόν για το θέμα που συζητάμε, αλλά απορρίπτω πλήρω τι εκκλήσει για περισσότερη εναρμόνιση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην απασχόληση. Οποιασδήποτε απόπειρε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό, να υπάρξει ένας ευρωπαϊκός ελάχιστος μισθός, οποιασδήποτε εκκλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει ελέγχους και κυρώσεις για τις εθνικές αγορές εργασίας, τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά σχέδια για τη δράση δεν δημιουργούν θέσεις εργασία. Οι επιχειρήσει, οι επιχειρηματίε δημιουργούν θέσεις εργασία. Δεν πρέπει να εισαγάγουμε μέτρα που να έχουν ε, αθέλητες παρενέργειες, που θα σταματάνε τους επιχειρηματίες, θα εμποδίζουν και τους αυτοπασχολούμενους να ε, λειτουργούν και να χορηγούν ενδεχόμενα και σε άλλους θέσει εργασίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις αυτή τη στιγμή ε, έχουν 19 εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τεράστιο δυναμικό για περαιτέρω ανάπτυξη, περαιτέρω θέσεις εργασία καινοτομία. Πρέπει να τις βοηθήσουμε, όχι να τις εμποδίζουμε. Ευρώπη τη Ελευθερία και Δημοκρατίας. Ε, το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Χέλμερ για 1,5 λεπτό. Ε, Mr. President, during the Second World War... Κύριε Πρόεδρε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η βασιλική αεροπορία ανησυχούσε για τις απώλειες των βαρέων βομβαρδιστικών. Οπότε προστάτευε τα πληρώματα της πρώτα απ' όλα με θωράκιση γύρω από τον πιλότο και μετά θωράκιση γύρω από τον ε, ναυτίλο κτλ. κτλ. Και όμως οι απώλειες ανέβαιναν και ανακάλυψαν πως είχε τόσο πολύ βάρος το αεροπλάνο που δεν μπορούσε να πετάξει καλά-καλά. Οπότε αφαίρεσαν όλη αυτή τη θωράκιση. Τα αεροπλάνα πετούσαν ψηλότερα και γρηγορότερα και οι απώλειες μειώθηκαν. Κύριε Πρόεδρε, εδώ και δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση φορτώνει κανονισμούς στην αγορά εργασίας με τις καλύτερες προθέσεις για να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Αλλά το αποτέλεσμα είναι μια αγορά εργασίας τόσο παραφορτωμένη και ανελαστική ώστε δεν μπορεί να πετάξει και επιπλέον τώρα μιλάτε και για πράσινε δουλειέ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα έπρεπε να ξέρουν πώς υπάρχουν μελέτες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αξιόπιστες μελέτες που δείχνουν πω υπαρχουν δουλειά κοστίζει απο θέσει εργασία στην πραγματική οικονομία, γιατί είναι τόσο ακριβή η πράσινη ενέργεια που δειχνουν πω καθε κοστίζει 2, 3, 4 θεσει εργασια στην πραγματική οικονομία γιατί είναι τόσο ακριβή η πράσινη ενέργεια που περιορίζει την ανάπτυξη στην υπόλοιπη οικονομία. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι πρώτα απ' όλα απορρίθμιση και δεύτερον να εγκαταλείψουμε τις πράσινες φιλοδοξίες μας. Εξ ονόματος της ε, Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτική Αριστεράς, Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Ινές Κριστίνα Ζούμπερ. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το, αυτή η δέσμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει και άλλα μέτρα, μείωση του φόρτου του κεφαλαίου, ενώ επιβαρύνει τους εργαζόμενους. Ε, δηλαδή υπερασπίζεται τη μείωση του κόστους της εργασίας, την αποκεφαλαιοποίηση των, ε, των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, την ιδιωτικοποίηση των συστημάτων αυτών και τρομοκρατεί τους εργαζόμενους. Εσείς θέλετε να μπορούν να μεταφερθούν οι εταιρείε. Μα πού να πάνε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει όλα αυτά η υποκατάσταση των δημοσίων υπηρεσιών μετατρέποντας τα δικαιώματα των εργαζομένων ε, η Κομισιόν θέλει να ορίσει και τους μισθούς με βάση την παραγωγικότητα, έτσι ώστε πάνω στους εργαζόμενους να φορτώσει την ευθύνη των, ε, της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Αυτό το πακέτο θέλει να αυξήσει την ευελιξία των εργαζομένων, την αύξηση των ωραρίων και τη δυνατότητα κινητικότητα των εργαζομένων, δηλαδή προωθεί την μετανάστευση λόγω έλλειψης ε, απασχόλησης. Θέλει να προωθήσει, λέει, δίθεν την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ενώ η ίδια καταργεί ένα σωρό θέσει απασχόληση μέσω των μέτρων. Πρέπει να πάψει αυτή την ε, δημαγωγία η Κομισιόν. Θέλουμε, απαιτούμε το τέλος των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μέσω των επενδύσεων στο δημόσιο τομέα και μέσω της αύξησης των μισθών. Ευχαριστώ. Οι άλλοι εγγεγραμμένοι ομιλητές, ε, το βήμα τον συνάδελφο κύριο Τόμας Μαν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λόγω της διαρκούς κρίσης έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ανεργία και τα κράτη-μέλη επιδίδεται το ένα στο άλλο. Πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Χρειαζόμαστε ειδικά ε, προσαρμοσμένες λύσεις για κάθε περιοχή. Πρέπει να βελτιώσουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πράσινες εργασίες, να αναγνωρίζουμε τα διπλώματα αμοιβαία, να αξιοποιούμε τα περιφερειακά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και όλα τα άλλα μέσα. Χρειαζόμαστε περισσότερη ελαστικότητα για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίες, αλλά και για να διασφαλίσουμε τις σταθερές θέσεις εργασίες. Πρέπει να απογορευτεί η μαύρη εργασία. Πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι αυτό θα δώσει και περισσότερα έσοδα στου προπολογισμού. Οι ασταθεί θέσει εργασία και οι μισθοί dumping πρέπει να απαγορευτούν να υπάρξει μια δίκαια αμοιβή. Οι συμφωνίε για μια ε, ελάχιστη αμοιβή είναι θέμα των κοινωνικών εταίρων. Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Πρέπει να υπάρξει εγγύηση για τους νέους. Μετά τέσσερις μήνες ανεργία πρέπει οπωσδήποτε είτε θέσει μαθητείας για επιπλέον ε, εξειδίκευση ή θέση εργασίας. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Αλλά οι επενδύσεις δεν πρέπει να προκύψουν από νέο, νέο δανεισμό μέσω ε, μεταρρυθμίσεων στις, ε, στα κράτη-μέλη και ισοσχελισμένων προϋπολογισμών θα έχουμε την ε, αναγκαία ανάπτυξη. Έτσι θα κάνουμε τις επιθυμίες μας, όχι απλώς επιθυμίες, αλλά πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Επιτέλους, ακούμε κάτι το έξυπνο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα υπάρξει ανάκαμψη αν η στρατηγική μας δεν δημιουργήσει τέσσερις εργασίες. Ευχαριστώ που ανοίγει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ για το σχέδιο δράση. Θα σα στηρίξουμε. Αλλά κύριε Επίτροπε, δεν επαρκεί η ανακοίνωσή σα. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για να αντιμετωπιστεί με τα μέτρα που λέτε. Πολύ σύντομα. Δύο σχόλια. Το πρώτο, η ανακοίνωση πρέπει να καταργήσει τις αντιφάσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών. Δεν είναι δυνατόν να ζητάτε, όπως δίκαια λέγεται, να επαναξιοποιούνται οι πόροι, ενώ στην ουσία δεν έχετε πόρους. Διότι υπάρχουν άλλες πολιτικές της Ένωσης που εμποδίζουν να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά για την κατάρτιση ή για δημιουργικές επενδύσεις. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε υπέρ μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασία που καταστρέφουν την απασχόληση. Και κύριε Επίτροπε, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ευρωπαϊκή εγγύηση για του νέου. Ευρωπαία. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτά που έχουν τι περισσότερε δυσχέρειε δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εκατό δισεκατομμύρια δώσαμε στη χώρα μου για πέντε τράπεζε. Δώστε 10 δισεκατομμύρια για να σώσουμε 5 εκατομμύρια νέου από την ανεργία. Αυτό θα ήταν ρεαλιστική δράση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Μάριαν Χάρκιν. Για ένα λεπτό. Thank you, Mr. Chairman. Towards job... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το να μιλάμε για ανάκαμψη με αυτές τις θέσεις απασχόλησης είναι πολύ εμπνευσμένο θέμα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η απασχόληση με τις κοινωνικές ανησυχίες να μην ε, βρίσκονται πίσω από τις οικονομικές ε, ανησυχίες. Ωραία λόγια, Καιρό τώρα να τα κάνουμε πραγματικότητα και να δώσουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Μια καλή πρόταση είναι η δημιουργία του ευρωπαϊκού επενδυτικού πακέτου, το οποίο θα αναλάβουν όλα τα κρατημέλη ώστε να δώσουν βιώσιμε θέσει απασχόληση. Το πακέτο αυτό θα έδινε ένα μήνυμα στου πολίτε ξεκάθαρο ότι σοβαρά προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τα μέτρα λιτότητα στην λιτότητα και την πειθαρχία με το σύμφωνο για την ε, ανάκαμψη και την απασχόληση. Ξέρω πως ε, μεγάλο ποσοστό των Ελλανδών υποψήφισαν την συνθήκη την δημοσιονομική, αλλά με πολλαπλές ελπίδες το έκαναν αυτό και ένα ε, μέσο για να το επιτύχουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό και κάνω έκκληση να μην εμποδίσετε τη συνέχισή του, να συνεργαστείτε ότι να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ε, προστιθέμενη αξία, αναβαθμίζοντας τους ε, ανέργους. για Monsieur le Commissaire, nous sommes... Κύριε Επίτροπε, Όλοι κάνουμε την ίδια διαπίστωση. Η κατάσταση τη απασχόληση στην Ευρώπη είναι καταστροφική. Εν τέταρτο των νέων κάτω των 25 ετών στην ανεργία τεράστια πρόκληση για τη νέα γενιά που αρνείται να είναι μια θυσιασμένη γενιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε το δρόμο με αυτό το πακέτο για την απασχόληση που στόχο έχει να δημιουργήσει 17 εκατομμύρια θέσεις μέχρι το 2020. Αλλά εξακολουθεί να μας ε, οδηγεί σε σύγκρουση. Καταδικάζει τους πιο ευάλωτους στις χειρότερες δυσκολίες. Ωστόσο, είναι εύκολο να βγούμε από την κρίση. Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή η οικολογική και κοινωνική μετατροπή τη οικονομία μα. Γι' αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν θέσει πράσινε, βιώσιμε, που δεν είναι δυνατόν να μετεκατασταθούν με συγκεκριμένε επενδύσει σε πράσινε καινοτόμε βιομηχανίε επενδύσεις στην ε, καινοτομία και στην, και στην μαθητεία διαβίου. Έπειτα αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης με λήψη υπόψη των ε, οδηγιών του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Είναι σημαντικό να ανυψωθεί και πάλι ο ελάχιστο μισθό για να τελειώσει το σκάνδαλο των φτωχών εργαζόμενων και για να καταπολεμηθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ. Έχουμε τα μέσα να σταματήσουμε αυτή την μάστιγα της ανεργίας. Είναι δυνατόν. Τι μας λείπει. Λείπει η πολιτική βούληση. Γι' αυτό είναι ευθύνη δική μας ε, όταν βλέπουμε ότι ο κύριος Μπαρόζο έβαλε πρώτη προτεραιότητα το θέμα της νεότητας και την ε, νεανική ενεργεία και τρία χρόνια μετά δεν έχουμε απολύτως τίποτα, καμία συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα είναι πήγουσα η κατάσταση πια και πρέπει να δράσουμε. Ο είναι ο συνάδελφος κύριος ε, Γιάτσεκ Βλόσοβιτς. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η στρατηγική Ευρώπη 2020 προϋποθέτει ότι 70% ε, σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να είναι σε πλήρη απασχόληση μέχρι το 2020. Στοχευμένη λοιπόν ανάπτυξη χρειάζεται. 17,5 εκατομμύρια έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση, Πολύ φιλόδοξο στόχο και για την Ένωση στο σύνολο αλλά και για την οικονομία των κρατών μελών ξεχωριστά. Η ενεργία ωστόσο αυξάνεται 9,5% το 2010, 10,2% το 2012. Συμπέρασμα. Έχουμε χάσει 6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης έκτοτε. Πού είναι η προοπτική για το πακέτο του κλίματος, ας πούμε, θα μπορούσαμε στη χώρα μου στην Πολωνία να ε, έχουμε αντί για δημιουργία θέσεων απασχόλησης απώλεια θέσεων εργασίας μέχρι μισό εκατομμύριο. Είναι καλή η στόχη και σημαντική, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε την αυτοαπασχόληση και καλείται επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ε, στις ε, διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και κρατικών προμηθειών. Η μείωση των κονδυλίων συνοχή δεν ξέρω μπορεί να, να είναι ηθική. Τόμας Χέντελ, για ένα λεπτό. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, εκτιμώ την πρότασή σας ε, για την παραγωγικότητα πάρα πολύ, αλλά αντί για το κατώτατο μισθό υποχωρήσατε απέναντι στην κυρία Μέρκελ και για τη δημιουργία θέσει απασχόληση στην υγεία δεν σας πιστεύω. Πώς θα δημιουργηθούν νέε θέσεις απασχόλησης αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα ανάγκασε τις χώρες του Νότου και της ε, Ανατολικής Ευρώπης να μειώσουν τις κλίνες στα νοσοκομεία μέχρι και στο μισό. Στις νέες χώρες δίνονται νέες συστάσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί ορισμένα κράτη-μέλη να μειώσουν ακόμα περισσότερο τις δαπάνες στην υγεία. Εγώ φοβούμαι ότι αυτά είναι εξαγγελίες και μόνο και όχι πραγματική ε, πρωτοβουλία για θέσεις απασχόλησης. Το αντίθετο. Σήμερα οικονομίε παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού λείπουν φάρμακα και υλικά νοσοκομιακά. σώνουμε συνέχεια τις τράπεζες. Πότε θα σώσουμε τους ανθρώπους και ιδιαίτερα την υγειονομική τους περίθαλψη σε χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση. Ευχαριστώ. Ε, επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Ντανούτα Γιαζοβέσκα. Για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον κύριο Βαρόσο στην παρουσίαση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό μου θυμίζουν κάτι που είχε πει ένας Αμερικάνος επενδυτής που έλεγε ότι ε, δεν δημιουργούν θέσεις απασχόλησης οι εργοδότες λέει αλλά οι καταναλωτές. Θα πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας και να ξέρουμε ότι πρέπει να τονωθεί η ζήτηση εσωτερική και εξωτερική. Να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν κίνητρα για την κατανάλωση και για ε, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Και κάποιες ε, άλλες μορφές εργασίας, άτυπες, όχι στάνταρ, θα πρέπει να εξεταστούν στην αγορά εργασίας έχουμε πολύ μεγάλο χάσμα σε ό,τι αφορά τα ε, δικαιώματα των εργαζομένων, ε, εξού και η φτώχεια και ο αποκλεισμός. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να έχουν ε, ασφάλεια εκτός από ευελιξία στην αγορά εργασίας και πάντα να λειτουργούμε προδιαγραφές και πρότυπα για την αμοιβή, για να μην έχουμε επισφαλείς μορφές εργασίας και νέες μορφές φτώχεια των εργαζομένων. Οι πολίτες θα πρέπει να κινητοποιηθούν και τα κράτη-μέλη να βρουν προληπτικά στις ε, συνθήκες οικονομίας που αλλάζουν συνεχώς. Προτεραιότητα επίσης έχουν και τα προβλήματα των νέων. επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επενδύσει στον τομέα της παιδείας και της επαγγελματικής κατάρτισης και ε, της απόκτησης ε, δεξιοτήτων. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει πολλές χρήσιμες προτάσεις. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει και σε συγκεκριμένα νομοθετικά βήματα. Ευχαριστώ. Την συνάδελφο κυρία Σιλβάνα Ράπτη για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, καλό το πακέτο της απασχόλησης, μόνο που πρέπει να φτάσει εγκαίρως στον παραλήπτη χάσαμε δύο ολόκληρα χρόνια φωνάζαμε συνεχώς εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ότι κάτι πρέπει να γίνει για την απασχόληση. αν χάσουμε άλλα δύο χρόνια μέχρι να εφαρμοστούν τα όσα λέγονται και τα όσα γράφονται φοβάμαι ότι θα είναι αργά. δεύτερο ζήτημα η αγορά εργασίας να είμαστε ειλικρινείς πλήττεται γιατί απέτυχαν οι μακροοικονομικές πολιτικές και έχουμε τώρα την κρίση αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας γιατί σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο μόνο μέσα στο 2011 έντεκα ο αντίκτυπος της κρίσης ήταν δραματικός. μερικοί απλοί αριθμοί ένας στους πέντε ευρωπαίους ένας στους δύο έλληνες φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του. δεύτεροι αριθμοί πέντε στους δέκα ευρωπαίους οχτώ στους δέκα έλληνες φοβούνται ότι αν χάσουν τη δουλειά τους δεν πρόκειται να βρουν άλλη θέση εργασίας μέσα σε έξι μήνες. αυτή είναι η πραγματικότητα και έρχομαι λοιπόν και σας καλώ το θέμα της ελαστικότητας το θέμα της ευελιξίας να το σκεφτόμαστε όχι μόνο σε σχέση με την εργασία να το σκεφτόμαστε και σε σχέση με την διάθεση των κονδυλίων και επειδή μιλάμε συνεχώ και για το θέμα τη ανταγωνιστικότητα, πρέπει να το καταλάβουμε μια και καλή πρώτον η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να είναι ένα θέμα που αφορά κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά είναι υπόθεση ολόκληρης της ευρωπαϊκής ένωσης αν θέλουμε δυνατή ευρωπαϊκή ένωση δυνατό ευρώ. γι' αυτό λοιπόν εάν από τη μια μεριά μονίμως ακούμε για μείωση των μισθών για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα σε κάποια κράτη μέλη εγώ θα έλεγα και το εξή γιατί να μην αυξηθούν στη γερμανία για παράδειγμα οι μισθοί ώστε να βοηθηθούν στην ανταγωνιστικότητά του τα άλλα κράτη που υποφέρουν. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ράπτη. Ε, επόμενος είναι ο συνάδελφος κύριος Γιάροσλαβ Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η οικονομία βρίσκεται σε μια στασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μας αναγκάζει να προβληματιστούμε για το πώς θα τονωθεί η ανάπτυξη και η μεγέθυνση της οικονομίας. Κατανοώ τα μέτρα εξυγίανσης των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παραβλέπει ορισμένες αιτίες αυτής της στασιμότητας της οικονομίας οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη χάνουν ε, τις δουλειές τους διότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες απλούστατα μετεγκαθίσταται. Φεύγουν από την Ευρώπη. Κοιτάξτε τι γίνεται στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στην Κίνα παράγονται τώρα τα αυτοκίνητα, στη Βραζιλία, στη Ρωσία και αλλού ανά τον κόσμο. Οπότε δεν είναι απορία άξιων ότι στην Ευρώπη ε, μειώνονται οι πωλήσει αυτοκινήτων σε σχέση με το παρελθόν. Τα εισοδήματα δεν είναι στην Ευρώπη, ούτε στους δικούς μας φορολογικούς ε, κορβανάδες. Έχουμε προβληματιστεί κύριε Επίτροπε τι θα γίνει στην Ευρώπη αν φύγουν σιγά σιγά όλοι. Ε, Κύριος Πατρίκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, υπάρχει μια βασική αντίφαση στις ε, επιλογές σας. Συνδέεται ε, την ε, χρηματοοικονομική εποπτεία με τη μείωση της κατανάλωσης των πολιτών. Ικανοποιούνται οι τράπεζες και αυτό ε, είναι σαν να προσπαθείτε να παντρέψετε το νερό με τη φωτιά. Δεν γίνεται. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα έρθει η ανάκαμψη. Ε, μειώνεται συνεχώς ο πλούτος που παράγεται. Η ανάπτυξη της εργασίας και της απασχόλησης δεν μπορεί να γίνει παρά με νέα κατανομή του πλούτου. Δηλαδή καλύτερη αμοιβή για την εργασία και καλύτερη αμοιβή για τις συντάξεις. Ε, και ένας νέος τρόπος να παράγεται πλούτος με την οικολογική μετάβαση της παραγωγής που θα δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη. Από την άλλη θα πρέπει να αντικατασταθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας που είναι μηχανισμός λιτότητας σε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο που θα συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα δίνει ε, νέο δάνειο που θα συνδέεται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την κατάρτιση, την οικολογική πρόοδο και ε, προωθώντας τα δημόσια αγαθά και τις δημόσια δημόσιες υπηρεσίες, στο νερό, στην ενέργεια, τις μεταφορές, την υγεία, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την παιδεία και τον πολιτισμό. Αλλιώς δεν θα γίνουν αυτά που τάζετε. Δίνω τώρα το λόγο στη συνάδελφο κυρία Ρεζίνα Μπαστός για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Από το 2008 η Ευρώπη έχει χάσει πάνω από εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Στη δική μου χώρα, την Πορτογαλία, η οικονομία ε, υποφέρει, επιβραδύνεται ε, με καταστάσεις πρωτόγνωρες. Ε, η ανεργία των νέων, των γυναικών φτάνει στα ιστορικά επίπεδα. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί επιπλέον την επόμενη διετία στα πλαίσια αυτά χαιρόμαστε βεβαίως για το νέο πακέτο για την απασχόληση και συγχαίρουμε τον Επίτροπο Άντορ. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην ανάγκη μεγέθηση της οικονομίας και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης νέες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν αν μειωθεί η φορολόγηση της εργασίας, αν ε, δημιουργηθούν, συσταθούν νέες εταιρείες, ε, ενισχυθούν ε, νέοι επιχειρηματίες, μικρομεσαίες κτλ. Οι εθνικές πολιτικές απασχόλησης θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι όπου δημιουργούνται περισσότερες θέσεις ε, εργασίας και ε, όπου υπάρχει χώρος είναι η τεχνολογία, η εκπαίδευση, η υγεία και η πράσινη οικονομία. Εκεί θα δημιουργηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα ε, στις δεξιότητες που ζητάει η αγορά και εκείνες που παρέχει η εκπαίδευση για να καταπολεμήσουμε την ανεργία θα πρέπει να έχουμε και κινητικότητα των εργαζομένων. Είναι απολύτως απαραίτητο επίσης να χρησιμοποιούμε τα διαρθρωτικά ταμεία προς την κατεύθυνση αυτή και αυτό είναι το κατεξοχή μέσο για να μπορέσουμε να δώσουμε νέες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Η κοινωνική διακυβέρνηση πρέπει να ε, ευνοηθεί επίσης διότι οι πολίτες μας περιμένουν αποτελέσματα από εμάς συγκεκριμένα. Ο ομιλητής είναι ο κύριος Ήμερ. Κώστελο για ένα... η κυρία συγγνώμη, Ήμερ Κώστελο για ένα λεπτό. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ένα από τα βασικά ε, μηνύματα του ε, δημοψηφίσματος ε, της Ιρλανδίας είναι ότι η απασχόληση είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα υπέρ της ατζέντα ανάπτυξης. Πρέπει να υπάρξει επίσης ε, βελτίωση, ένα πρόγραμμα το οποίο θα σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, να προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη, να αντιμετωπίζει ε, την φτώχεια και το κοινωνικό dumping, να προστατεύονται οι ευάλωτοι, οι μερική απασχόληση και όλοι εκείνοι που είναι παγιδευμένοι στη μαύρη οικονομία. Ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει την ανάγκη επενδύσεων ε, και θα πρέπει να διατίθενται τα κονδύλια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι είναι η ραχοκοκαλιά τη οικονομία. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένε πράξει για να αντιμετωπιστεί η ενεργεία των νέων, ε, να υπάρχουν ευρωπαϊκέ εγγύσει, να προσαρμοστεί επίση ε, και η ποιότητα ε, σε στάζ πολλοί βρίσκονται σε τέτοια διαδικασία χωρίς καμία προοπτική απασχόληση. Εμείς λοιπόν χαιρετίζουμε τη δική σας πρόταση και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Σας ευχαριστώ. Ε, διαδέχεται στο βήμα η συνάδελφος κυρία Βερόνικα Λόπε Φοντανέ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πακέτο της απασχόλησης. Φιλόδοξος ο στόχος και πρόκληση στα πλαίσια της σημερινής κρίσης. Θα πρέπει όμως να καταφέρουμε να επιτύχουμε τη στρατηγική του 2020 και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο είναι απαραίτητο να μεταρρυθμίσουμε τις αγορές εργασίας για να είναι πιο δυναμικές και πιο ε, πρόσφορες στο να ε, εργάζονται ε, οι άνθρωποι και να μην χάνουν τη δουλειά τους όταν γίνονται διαρθωτικές προσαρμογές να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης όχι μόνο σε περιόδους ε, ανάκαμψης της οικονομίας. Η φορολογία θα πρέπει να είναι αντίστοιχη, να ε, δίνει κίνητρα για την πρόσληψη υπαλλήλων, να δίνει κίνητρα για την αυταπασχόληση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε νέες επιχειρήσεις. Βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας ε, των πιο ευάλωτων ομάδων που είναι οι γυναίκες και οι νέοι και επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις άτυπες ε, ή άδειλες ε, μορφές εργασίας. Είναι σημαντικό αυτό γιατί παρόλο που είναι πολύ ψηλή η ανεργία, που ειναι η ανεργια ολο και περισσότερο θέσεις απασχόλησης υφιστάμενες δεν καλύπτονται γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό με τα προσόντα που ζητούν. Θα πρέπει να καλυφθεί αυτό. Χρειάζεται περισσότερη δυνατότητα και ευελιξία και γεωγραφική κινητικότητα. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να προχωρήσουμε με στένος αποφασισμένοι για τη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας πανευρωπαϊκής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ε, επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος κύριος Σέρτζιο Γκαϊτάνο Κοφεράτη για ένα λεπτό. Grazie, Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ πιστεύω ότι έχουμε δύο στόχους που πρέπει να επιδιώξουμε για να τους υλοποιήσουμε. Ο πρώτος αφορά την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Γνωρίζουμε ότι η προτεραιότητα είναι να ασχοληθούμε με τους νέους και γνωρίζουμε ότι το σημαντικότερο εργαλείο είναι η εκπαίδευση. Ότι επενδύει κανεί στην εκπαίδευση ε, θα αποδώσει στην ανάπτυξη και στην ε, κοινωνία. Ε, βέβαια δυστυχώς γι' αυτό μιλάμε λιγότερο. Μιλάμε ε, λιγότερο για τη ρύθμιση της μαύρης ε, εργασίας. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, που εργάζονται χωρίς συμβάσεις, χωρίς να αναγνωρίζονται τα εργατικά τους δικαιώματα, αλλά ούτε και το δικαίωμα στην ηθαγένεια. Γιατί πολύ συχνά είναι άτομα που έρχονται σε εμά χωρίς να έχουν άδεια παραμονής και τις ίδιες συνθήκες όπως οι άλλοι. Πρόκειται λοιπόν για πραγματική εκμετάλλευση, αλλά πρόκειται και για ουσιαστική στρέβλωση Τη αγορά εργασία. Γι' αυτό λοιπόν αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα να τους δώσουμε την ίδια σημασία, δηλαδή τέσσερις εργασίες για τους νέους, αλλά και παράλληλα να ρυθμίσουμε αυτό που ήδη υπάρχει και δυστυχώς δεν ε, ρυθμίζεται από νομοθεσία. Κύριος Κωνσταντίνος Πουπάκης για δύο λεπτά. Πρόεδρε κύριε Πέτροπε, η ανεργία αποτελεί ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρόβλημα με οδυνηρές επιπτώσεις για την κοινωνική συνοχή και την πραγματική οικονομία της ένωσης. σε κάθε νέα μέτρησή της σημειώνει ιστορικό υψηλό για πολλές ευρωπαϊκές χώρες και το 45% των ευρωπαίων πολιτών σύμφωνα με το τελευταίο ευρωμαρόμετρο ανησυχεί για το έλλειμμα απασχόλησης. η ευρωπαϊκή ένωση δηλαδή βρίσκεται μπροστά σε μια κορυφαία πρόκληση με την απασχόληση να βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. είναι σαφές πω η αιμονή στι συνταγέ τη ακραία λιτότητα σε ορισμένε χώρε έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αύξηση τη ανεργία. στη χώρα μου την ελλάδα ήδη ένα στου τέσσερι πολίτε είναι εκτό αγορά εργασία με τη μακροχρόνια ανεργία να ξεπερνά το 55% και την ανεργία των νέων να αγγίζει το 53% καταδικάζοντα στην αδράνεια ή τη μετανάστευση το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία. ταυτόχρονα η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων όχι μόνο δεν συνέβαλε στη συγκράτηση απασχόλησης αλλά αντίθετα ανακύκλωσε φτώχεια και ύφεση. επιβάλλεται λοιπόν συνολικότερα να οθεί αναπτυξιακό περιεχόμενο στην οικονομική διακυβέρνηση γιατί δεν μπορεί η οικονομική βιωσιμότητα να αναζητείται αποκομμένη από το σφιγμό της κοινωνίας. άλλωστε τα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης συνιστούν σημαντικές κοινωνικές επενδύσεις. τέλος θα ήθελα να επισημάνω ότι κράτη μέλη όπως η ελλάδα που στηρίζονται οικονομικά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείονται από τη διαδικασία για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής. 2020. πρέπει λοιπόν να ακολουθεί ένα μείγμα πολιτικής που θα διασφαλίζει τη δημοσιονομική εξυγίανση θέτοντας παράλληλα τη βάση για μια αναπτυξιακή πορεία με νέε βιώσιμε και ποιοτικέ θέσει εργασία. και αυτό το ξέρετε πολύ καλά εσείς κύριε επίτροπε με την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχετε το ξέρετε πολύ καλά και εσεί κύριε πρόεδρε γιατί είσαστε πάντα κοντά στην κοινωνία και τα προβλήματά τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπάκη. Ε, επόμενη ομιλήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Κίνγκα Γκέντς. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπουμε ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με την ε, ανεργία, κυρίως για κάποιες κοινωνικές ομάδες που έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση ε, όπως ε, τα παιδιά, οι ανάπηροι, όσοι είναι ανάμεσα στα 50 και τα 55, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα νέο σχέδιο. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις της κρίσης, ε, κυρίως ε, σε κάποια πληθυσμιακά ε, στρώματα Οφείλουμε να απλουστεύσουμε το σύστημα, να προσφέρουμε ευκαιρίε επιμόρφωση, κατά τη επιμόρφωση και απασχόληση, ε, για να καταπολεμήσουμε αυτέ τι δυσλειτουργίε. Για να επιτύχουμε το στόχο μα, ε, θα έπρεπε ε, να διευκολύνουμε την καταβολή πληρωμών από τα συστήματα κοινωνική ασφάλιση, να βελτιώσουμε τη λειτουργία τη αγορά εργασία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην κρίση. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος ε, Χάιντς Μπέκα για 1,5 λεπτό. Κύριε Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση των Σημερινών Προκλήσεων, το σχέδιο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών ή με την ε, αύξηση των θέσεων εργασία. Όπω προσπαθούν να μα πείσουν διάφοροι λαϊκιστέ. Προφανώ, η ευθύνη η δική μα είναι να επιτύχουμε και του δύο στόχου. Υπάρχει μια δήλωση τη Κομισιόν ε, και αυτή η δήλωση είναι ένα σημαντικό βήμα προ τα εμπρό. Χαίρομαι πάρα πολύ ε, που αναγνωρίζεται την ικανότητα που έχει η οικονομία, το δυναμικό της, το διτό διοικό σύστημα εκπαίδευσης. Ε, χαίρομαι που οι τέσσερις μήνες της εγγύησης για τους νέους θα γίνει πραγματικότητα, ότι η διαβίου μάθηση ε, είναι σημαντική όλο και περισσότερο για τους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους και επίσης και ότι θα πρέπει να ορίζεται ακριβώς το ποια είναι τα μέτρα και μέσα που υπάρχουν. Τώρα λοιπόν τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί πρέπει να εφαρμοστούν από όλες τις δηλώσεις Κομισιόν ε, προκύπτει κάτι τέτοιο. Ε, να πω και κάτι για τον ε, δικαιολογημένο στόχο που είναι να μην χαθεί μια ολόκληρη γενιά. Όμως αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο μέσα από την εφαρμογή της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης ανάμεσα στις γενιές. Και αυτό προφανώς ξεκινάει με την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προβλήματων της σημερινής εποχής που είναι η εργασία. Αυτομάτως όμως οδηγεί ε, στο να μην υπάρχουν ε, χρέη. Εδώ λοιπόν δεν θα ήθελα να ε, τσακωνόμαστε αλλά να προσπαθήσουμε να ελοποιήσουμε και τους δύο στόχους. Αυτός πρέπει να είναι εξάλλου και ο σημαντικότερος στόχος του Κοινοβουλίου. Δεν βλέπω στην αίθουσα τη συνάδελφο κυρία Ματέρα και επομένως ε, εκείνη η διαδικασία catch the eye

Το, κύριε Πρόεδρε, οι νέες θέσεις υπάρχουν στο μυαλό μας, υπάρχουν στις απόψεις όλων αυτών των νέων που προσπαθούν να αυτοπροσδιοριστούν στην αγορά εργασίας. Ε, πολλοί δεν ξέρουν πώς πρέπει να τα κάνουν όλα αυτά. Οι ευκαιρίες για την απασχόληση μπορούν να αναζητηθούν στις υποστηρικτικές εργασίες για την υγεία των ανθρώπων. Ακριβώς όπως το συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μια ομάδα νέων στην ε, Σλοβενία ε, έχει προσφέρει ένα εργαλείο για τους τυφλούς έτσι ώστε να μπορούν οι τυφλοί αυτοί να αντιμετωπίζουν την καθημερινή του ζωή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινή του ζωή. Η αγορά για τους ανθρώπους με αναπηρία και αντιμετώπιση των αναγκών τους είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι συμφωνούμε ότι το μέλλον ανήκει στη νέα γενιά. Δυστυχώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νεολαία εκτέθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από όλους στην κρίση. Είναι λίγα ανησυχητική η κατάσταση και ως εκ τούτου κρίνω ότι αμελήτη οφείλουμε να αναλάβουμε μέτρα για να αναβαθμίσουμε την ζωή τους σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Θα Απευθύνω έκκληση λοιπόν προς τα κράτη-μέλη να προσδώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτήν την ε, κατηγορία του πληθυσμού και στα εθνικά στρατηγικά προγράμματά τους να συμπεριλάβουν ε, ε, την κατάλληλη πρόσβαση για τους νέους ε, στην αγορά εργασίας, καθώς και να προσφέρουν ε, δυνατότητες απασχόλησης αλλά και κατάρτισης. Πιστεύω ότι αυτό χρειαζόμαστε, ούτως ώστε μια γενιά να ζήσει σε ένα ασφαλής μέλλον. Η κυρία Ελίζαμπετ Σρόιντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαιρετίζω το γεγονός ότι στο σύμφωνο απασχόλησης ε, την ε, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την υιοθετήσατε. Λέτε ε, στην έκθεσή σας ε, ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας μετά το 2020. Αυτό είναι δυνατόν, είναι πιθανό, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να οριοθετήσει το βιομηχανικό πολιτικό πλαίσιο και μάλιστα ως μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Ε, πιο συγκεκριμένα αυτό σημαίνει το εξή. Αν δεν υπάρχει μία φιλόδοξη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, δεν θα υπάρχει και ανάγκη για εργαζόμενους στον οικοδομικό τομέα. Δηλαδή εσείς ε, οφείλετε να βρείτε τη λύση μαζί με τους συναδέλφους σας έτσι ώστε να οριοθετήσουμε πολιτικά αυτό το θέμα. Γιατί αλλιώς σας το λέω ευθύς εκ των αυτά τα οποία είπατε δεν θα υλοποιηθούν και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε στον εαυτό μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε και την αξιοπιστία της Ένωσης αυτής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση είναι το βασικό μέσο να λυθούν τα πιο ξεά προβλήματα στην Ευρώπη, που είναι η φτώχεια και η ενεργεία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Ε, μόνο έτσι θα επιστρέψουμε στο δρόμο της ανάπτυξης. Πρέπει να επενδύσουμε στην επιχειρηματικότητα και να καταργήσουμε τη γραφειοκρατία και τους νομοθετικούς φραγμούς που μπλοκάρουν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 70% των θέσεων απασχόληση είναι στις μικρομεσαίες. Επίσης, ε, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και της ε, εργασίας. Είναι μεγάλη ενεργία και παρόλα αυτά δεν καλύπτονται και νέες θέσεις εργασίας οι νέοι μας μπορεί να είναι μορφωμένοι, αλλά δεν είναι σωστά καταρτισμένοι για να ε, είναι και απασχολήσιμοι, όπως λέγεται, σε θέσεις που ζητούν οι επιχειρήσεις. Χρειάζονται νέες λύσεις παντού. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κυρία Εύελιν Ρέγνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Να κάνω μια παρατήρηση, αν επιτρέπετε, μετά τη συζήτηση εδώ στην αίθουσα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι γεμάτη η αίθουσα. Το αξίζει και το θέμα και είναι νέοι στην Ευρώπη. Στη συνθήκη τη Ευρωπαϊκής Ένωση έχουμε στόχο για την απασχόληση, έχουμε τόσε πολλές προποθέσει που είναι δεδομένες και το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Γι' αυτό παρατηρώ το εξή. Την περασμένη φορά στη συζήτηση τη Αλομέλειας για την ανεργία των νέων είπατε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, ταιριάζει και στο σημερινό θέμα. Δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ε, την σύνολη εικόνα προφθαλμού να έχουμε μια μακροοικονομική πολιτική στραμμένη προς την απασχόληση. Αλλιώς δεν πρόκειται να λυθεί μόνο με μέτρα απασχόλησης αυτό το θέμα της ανεργίας. Χρειάζεται οικονομική πολιτική και ιδιαίτερα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να ε, δώσουμε εκείνα τα χρήματα που χρειάζονται οι άνεργοι στην Ευρώπη και αξίζουν. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch the Eye και τώρα δίνω το λόγο τον Επίτροπο κύριο Άντορ Λάσλο Άντορ. You Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές ε, για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και απευθύνει σαφέστατα μηνύματα προς την Επιτροπή σχετικά με το πακέτο απασχόλησης και τη μελλοντική πορεία μας. Δεν χρειαζόμαστε μόνο καλά έγγραφα, πρέπει να φροντίσουμε ούτως ώστε να είναι σωστή η εφαρμογή και γι' αυτό πραγματευόμαστε όλα αυτά ε, τα ζητήματα. Γνωρίζετε σίγουρα τη δράση που έχουμε αναλάβει από πλευρά τη Επιτροπή αλλά και τι ευρύτερε πολιτικέ απασχόλεις. Την επόμενη εβδομάδα ε, θα συναντηθούμε στα πλαίσια τη ομάδα εργασία των κοινωνικών εταίρων, επιδιώκοντα ε, μεγαλύτερη συνεργασία για τι επιμέρου πτυχέ του πακέτου απασχόληση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω την ε, σημασία πολλών παρατηρήσεων ως προς το ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής απασχόλησης ε, διότι δεν μπορείτε να αποκόψετε την απασχόληση ε, από το ευρύτερο οικονομικό τοπίο. Ένα τρίτο της ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επίπτωση απόρρια της κρίσης και σε κάποια κράτη-μέλη ε, αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο ίμιση ή και περισσότερο. Χρειαζόμαστε αυτά αποτελέσματα, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ε, ε, έχουμε κατά νου την κρίση και θέλουμε η οικονομία να αντεπεξέλθει στην κρίση. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα χειριστούμε το δημόσιο χρέο και το χρέο του ιδιωτικού τομέα. Με το που βρούμε τις πλέον πρόσφορες λύσεις ε, για όλα αυτά τα ζητήματα θα βελτιωθεί και το μακροοικονομικό ε, περιβάλλον και θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε ενεργείστερα με τις πολιτικές απασχόλησεις. Ε, πέραν αυτού λοιπόν αληθεύει ότι χρειαζόμαστε καλύτερες λύσεις για να βοηθήσουμε τους ανέργους. Όταν σας μιλάω για το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο, είναι εξίσου σημαντικό να ασχοληθούμε με το ζήτημα των επενδύσεων και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας. Συμμερίζομαι τις απόψει κυρίας Χάρκιν για τη σημασία των επενδύσεων ή της βιομηχανικής πολιτικής η κυρία Σρέτερ και ο κύριος ε, Πάσκο μου απίθυναν ερωτήσεις ε, και όντως ασχολούμαστε ε, επισταμένα με την ε, βιομηχανική πολιτική, κυρίως με τη διάσταση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η ικανότητα αναζωογονήσει ε, τη ε, βιομηχανία ε, για να δημιουργηθούν βιώσιμε θέσει απασχόλησης έχει κέρια σημασία. Το πακέτο απασχόλησης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως δομικό στοιχείο ενός νέου οικονομικού μοντέλου αν ε, ε, ε, πέρα από τους μισθούς, πέρα από τον νόμο της προσφοράς και ζήτησης που βλέπουμε στο πακέτο απασχόλησης, μπορώ να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Ο ρόλος οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Πιστεύω ότι αυτό μας ανοίγει νέα παράθυρα ευκαιρίες, η ικανότητα δηλαδή να εστιάσουμε την προσοχή μας σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα ζητήματα και με πιο αποτελεσματικό τρόπο, με στόχο πάντοτε την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ποιοτικών θέσεων απασχόληση. Δεν χρειάζεται τώρα να παριθμίσω όλους τους βουλευτές που παρενέβησαν, αλλά πολλοί από σας ε, τόνισαν ε, την ε, σημασία που έχουν είναι και θυμάστε την προηγούμενη συζήτησή μα. Ε, γίνονται πολλά πράγματα. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Ιταλία ε, και τα διαρθρωτικά ταμεία διαθέτουν ε, πάρα πολύ σημαντικά κονδύλια για να βοηθήσουν του νέου Στη Σικελία, μόνο να πάρουμε μία περιοχή, έχουμε φτάσει περίπου το μισό δίσε στα πλαίσια τη ανακατανομή των κονδυλίων και δεν είναι μόνο, για, είναι μόνο για αυτή την περιοχή, ούτε καν για ολόκληρη την Ιταλία. Ταυτόχρονα στα 8 ε, κράτη-μέλη όπου η ανεργία βρίσκεται σε, στα χειρότερα επίπεδα. Θα χρησιμοποιούμε επίσης την άσκηση της ανακατανομής. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης ε, το σύστημα των εγγυήσεων. Άκουσα τις απόψεις περί αυτού της κυρίας Μπερές και άλλων. Αυτά σε στεγνό συντονισμό με το Συμβούλιο θα αποφέρουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα προτού λήξει το τρέχον έτος και θα διαπιστώσουμε έτσι αν ε, κάποιες ε, ουσιαστικές ευεφάρμοστες ε, λύσεις θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Στα πλαίσια πάλι του πακέτου απασχόλησης θα παράγουμε την, το, το ποιοτικό πλαίσιο μετά το πέρα των διαβουλεύσεων που τώρα διεξάγονται με τους κοινωνικούς εταίρους. Για την μικροχρηματοδότηση και τι μικρομεσαίε επιχειρήσεις, οι κύριοι Μπένιον και Μάκεντάιρ τόνισαν επαρκώ τη σημασία του ζητήματος. Ε, ε όντως, ε, παραμελήσαμε λίγο τη σημασία αυτού, ε, μεταξύ άλλων, διότι η νέα γενιά ίσω δεν γνωρίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν σε χώρε όπως η Ιταλία. Χρησιμοποιήσω και πάλι αυτό το παράδειγμα, όπου υπήρχαν πολλές επιτυχημένε ιστορίες ε, ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, δεν υπάρχει λοιπόν μετάβαση προς τη νέα γενιά. Πάλι θέμα ανθρωπίνου κεφαλαίου, δηλαδή οι άνθρωποι οι ίδιοι θα ενισχύσουν τι γνώσει για την επιχείρηση και θα χρησιμοποιήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ούτω ώστε να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Στα πλαίσια πάλι των επιχειρήσεων, ε, πιστεύω δικαίω ε, η έμφαση στη σημασία των εταιριών κοινωνικού χαρακτήρα. Οι συνάδελφοι μίλησαν για την συμπερίληψη στην ε, κοινωνία κάποιων αποκλεισμένων ομάδων. Ο Επίτροπος Μπανιέ που μίλησε νωρίτερα συνεργάζεται στενά μαζί μου για αυτό το θέμα. Υπάρχουν και γενικέ διευθύνσει που συνεργάζονται με εκπροσώπου των κρατών μελών. Την περασμένη εβδομάδα, παραδείγματο χάρη, έγινε ένα σεμινάριο στι Βρυξέλλε όπου παρευρέθησαν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών με στόχο την προώθηση τη κοινωνική οικονομία στο ευρύτερο πλαίσιο σε όλα τα κράτη-μέλη. ούτω ώστε αυτέ οι ομάδε ε, που βρίσκονται σε δυσμενή θέση όπω οι ανάπηροι να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στην αγορά εργασία και στην κοινωνία. Ε, είτε μιλάμε για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, είτε μιλάμε για την κοινωνική οικονομία, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τη συζήτηση για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Ε, συνεχίζονται οι συζητήσει εδώ και στο Συμβούλιο για το επόμενο σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορεί μόνο να εστιάζουμε την προσοχή μα στην τωρινή ανακατανομία αλλά και στην ασφαλή χρηματοδότηση μέσω χρηματοπιστωτικών εργαλείων που μπορούν άμεσα να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει προεξέχουσα θέση από σε αυτό το πλαίσιο και πιστεύω ότι γνωρίζετε το περιεχόμενο της σχετικής πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την κυρία Χάρκιν σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Όντως ε, θα ήταν ιδιαίτερα προβληματικό να διακόψουμε την λειτουργία και τη στήριξη αυτού του ταμείου και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας ε, στον αγώνα που κάνουμε για να σώσουμε αυτό το ταμείο και να διατηρηθεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, έλαβα μία πρόταση ψηφίσματο για την περάτωση αυτή τη συζήτηση. Πέρα συζητήσεω, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στι 12 η ώρα. Τώρα εισάγεται προ συζήτηση η έκθεση του συναδέλφου κ. Γιάννο Όντερ με τίτλο Έλεγχο των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνε ουσίε. Θέση εισηγητή, καταλαμβάνει, θέση εισηγητού καταλαμβάνει ο συνάδελφος κύριος Ρίχαρτ Ζέιμπα